Συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσει η συνεδρίαση γιατί έχουμε και την ε, ψηφοφορία αλλά πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω αυτό το κατασκεύασμα εδώ μπροστά. Ο Τόμ Χάνκς και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Όχι εντάξει, απλά τραβάει εικόνες η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών για να συλλέξει εικόνες ε, για ένα ντοκιμαντέρ πανοραμικό 360 μοιρών που θα εξηγεί πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο εξού και όλες οι κάμερες. Τώρα, θα τραβάνε εικόνες ε, κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας ε, της έκθεσης Μαρινέσκου. Κύριε Μαρινέσκου θα γίνεται διάσημος και κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Επίτροπο τον κύριο Ταλιάνη. Οπότε χρειαζόμαστε πολλές κάμερες. Πρόκειται για ένα μέρος της γενικότερης ιδέας ε, του Γραφείου Επισκεπτών που ενέκρινε το Προεδρείο το 2008 για να δείξει τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επέλεξαν τρεις νομίζω ή τέσσερις μόνο επιτροπές. Τις σημαντικότερες ακριβώς για να τραβήξουν εικόνες. Γι' αυτό ήρθαν και σε επαφή ε, μαζί μου για να τράβηξουν κάποιες εικόνες από την Επιτροπή μας. Οπότε τυχαία θα τραβηχτούν κάποια πλάνα και κάποια πλάνα από την αυριανή Ολομέλεια. Οπότε υπάρχουν οι κανονικές κάμερες αλλά και αυτοί η θαυμάσια εδώ πέρα συσκευή μπροστά μου που μας δίνει την ε, πανοραμική εικόνα. Απλά σας ενημερώνω επειδή έχουμε ακριβώς πλάνα σε 360 μοίρες δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς ε, πουθενά. Δηλαδή αν βαξίνετε τη μύτη σας να έχετε κατά νου πως ε, σας ε, τραβάει η κάμερα για να μην δούμε συναδέλφους ε, να καταλήξουν στο μοντάζ αν θέλετε στο πάτωμα του μοντάζ λοιπόν αν ήξεραν πως θα φορέσει το καλό της καπελοκύρια Λιχτεμπέργκερ, θα είχαν άλλη κάμερα αλλά τέλος πάντων αυτές έχουμε. Οι κάμερες είναι εδώ πέρα λοιπόν από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας για να δει το κοινό πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο και είμαι σίγουρος πως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη ψηφοφορία της έκθεσης Μαρινέσκου για το φορά εμπορευματικών φορτίων με σιδηρόδρομο. Να υπενθυμίσω συναδέλφους πώς θα πρέπει να έχουν την κάρτα των ε, ψηφοφοριών και ξεκινάει τώρα μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Can we just make... Unfortunately, the Greens have gone in the wrong way. Yeah. Δυστυχώς, οι πράσινοι εκεί δεν τα κατάφεραν. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Okay, have we got no problems with... Ωραία, κανένα πρόβλημα με τα νούμερα. Όχι. Οπότε είμαστε έτοιμοι. This one. Πρώτα απ' όλα λοιπόν. Συμβαστική λύση Α καλύπτει τις τροπολογίες 12 και 96 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 14 του εισηγητή με προφορική τροπολογία που βλέπετε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 97 έχει αποσυρθεί, περνάμε στην 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 αποσύρεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 όχι καταπίπτει 105 του κυρίου Ρικέ επί του άρθρου 2 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 αποσύρεται συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Γ άρθρο 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 20 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή η 21 του εισηγητή με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα άρθρο 4 παράρτημα 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή άρθρο 7 παράγραφος 1 προφορική του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 με την προφορική τροπολογία της κυρίας Μπιλμπάου υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την 118 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 16 υπέρ, 17 κατά μια αποχή απορρίπτεται. 26 του συγητή με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ε, άρθρο 7 παράγραφος 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική σίγματα υπέρ κατά άποχες δεκτή 128 Λιμπεράτσκι με προφορική τροπολογία υπέρ κατά άποχες δεκτή Συμβαστική ζήτα άρθρο 7 παράγραφος 6α υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 του εισηγητή με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 8, παράγραφος 4, προφορική τροπολογία της κυρίας Μπιλμπάου. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 129 χωριστή ψηφοφορία που ζητάει ο κύριος Μαρινέσκου. Πρώτο μέρος μέχρι το Along with Other Measures. Το δεύτερο μέρος, it must also take into account, μέχρι Freak mary Μέρος πρώτο της 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τρίτο μέρος, να υπάρχει και τρίτο μέρος, τελευταία φράση της 129 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 33 του συγητή προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 34 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή άρθρο 10 παράγραφος 1 προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 35, 36, 37, 38 μέχρι το 42 έχουν αποσυρθεί ναι, εκτός, εκτός από τη 41. Ηρεμήστε. 41 υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 44 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 131 καταπίπτει, 45 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε λοιπόν τώρα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 12 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ κατά άποχες δεκτή συμβιβαστική ήττα στο 12α υπέρ κατά άποχες δεκτή 48 της υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά άποχες δεκτή 51 αποσύρεται 52 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά άποχες δεκτή 53 υπέρ κατά άποχες δεκτή 146 κυρίου Κράμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή Πενήντα έξι του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 148 και 149 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 57 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 διαγραφή υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 κατά πίπτη 64 του εισηγητή έχουμε περάσει το άρθρο 15 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 του κυρίου Κράμερ υπέρ κατά αποχές Α, απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές Α, απορρίπτεται 65 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 και 67 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 και 155 ταυτόσιμες κύριο Νερτούγκ και Τρεμόσα υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε τις 154 και 155 άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 ψήφισαν, 16 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στην 156 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 68 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 157-158 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές 159 καταπίπτει οπότε 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 20 παράγραφος 1 Τροπολογίες 70 έως 76 έχει προταθεί να ψηφιστούν αμπλοκ υπέρ κατά αποχές δεκτές. 77 αποσύρεται 78 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 160 κράμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κύριε Μαρινέσκου για την 161 ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αποσύρω την ε, προφορική τροπολογία και να ψηφιστεί αρχική 161. Ωραία, το καταλάβατε όλοι. Αποσύρεται η προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε επί της αρχικής. 161 η αρχική λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 162 υπέρ. Κατά. αποχής, δεκτή. 163 Μπιλμπάο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 164 με την προφορική τροπολογία γιατί υπήρχε κάποια σύγχυση που επανήλθε υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή 167 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 του εισηγητή έχει εγκριθεί μου λένε με τη συμβαστική δέλτα οπότε περνάμε στην 168 μια στιγμούλα Οπότε περνάμε στην 1. η 79 και 169 καταπίπτουν. Λοιπόν, εκτιμώντας 4 τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή Τέσσερα προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 τικάου υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 1 όχι θήτα υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 στο εκτιμώντας 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική γιώτα εκτιμώντας 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας 13.87 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται Έξι του εισηγητή με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 89 αποσύρονται Α, πρέπει να ψηφίσουμε στην 88 την δεύτερη φορά τον... εκεί που λέει σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη αναφορά των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην 88 αρχιτή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34 ψήφισαν, 22 υπέρ 12 κατά δεκτή. 7 και 89 καταπίπτουν. 90 Μαρκινιέβιτς υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 αποσύρεται. 91 Κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή είναι καταπίπτει 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 αποσύρεται 10 του εισηγητή προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 αποσύρεται 95 αποσύρεται νομίζω 95 της κυρίας Μπιλμπάου. Υπέρ. Όχι, όχι, ψηφίζουμε την 95, αυτό λέω. Γιατί η 11 έχει αποσυρθεί, πρέπει να ψηφίσουμε την 95 άρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. τελική ψηφοφορία. Εάν είστε έτοιμοι, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 36 ψήφισαν, 30 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Οπότε εγκρίνεται η έκθεση συγχαρητήρια στον κύριο Μαρινέσκο. Καλητήρια σε όλους. Αρκετά καλά τα πήγαμε. Τώρα έχουμε 10 ε, λεπτά μέχρι να έρθει ο Επίτροπος. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μην φύγετε για να ακούσετε τον ε, κύριο Ταγιάννη. Οπότε σε 10 λεπτά θα ξαναλέμε. Ευχαριστώ. Valeria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

Να ξαναρχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίαση και να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο Ταγιάννη. Ξέρουμε τον Επίτροπο. Θα το γνωρίζετε από τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές θητείες. Ήταν ε, μάλιστα Επίτροπος Μεταφορών πριν αναλάβει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Επίτροπε, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και περιμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε σχετικά με την πολιτική τουρισμού. Εγώ θα ακούσω πολύ προσεκτικά γιατί με ενδιαφέρουν ε, οι συντηρόδρομοι τα μάλα και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να σας ακούσουν με ανυπομονησία. Σας ευχαριστώ που προσφερθήκατε να έρθετε σήμερα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Ας μιλήσω Ιταλικά. Υπάρχει μια νομική βάση για τον τουρισμό στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, τα καταφέραμε γιατί δεν θέλω να εγκαταλείψω και τη σχέση μου με αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Χάρη λοιπόν στη συνθήκη της Λισαβόνας μπορώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου επί δύο χρόνια σχεδόν ε, καταφέραμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα και να στείλουμε καλά μηνύματα στους Ευρωπαίους ε, πολίτες και ελπίζω αυτό είναι ένα προμήνυμα για ότι θα συμβεί και σε αυτόν τον τομέα, τον τουρισμό, που για πρώτη φορά έχει νομική βάση. Και είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος Επίτροπος που έχει την ευθύνη για τον τουρισμό, με συγκεκριμένη νομική βάση. Χαίρομαι λοιπόν που αυτή την ευθύνη τη μοιράζομαι με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και με τον, Επίτροπο, και με τον Πρόεδρο της, τον κύριο Σίμψον. Στην Ένωση αναγνωρίζονται αρμοδιότητες με σκοπό να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων και να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Είναι μια πραγματική οριζόντια πολιτική. Τώρα, από κοινού θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την πολιτική. Σας ζητώ επίσημα να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια συνένεση και να καθορίσουμε το περιεχόμενο και να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για την πολιτική αυτή. Δεν μπορούμε να μείνουμε αναδρανείς απέναντι στον τουρισμό, που είναι ένα τουρισμό που είναι η τρίτη οικονομική δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρώπη εν γέννη. Τόσο σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, όσο και σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει. Πιστεύω, πιστεύω ότι είναι πραγματικά στρατηγική ε, στρατηγικό τομέα ε, για την οικονομία χάρη στην ε, ικανότητα για ανάπτυξη και απασχόληση. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι αποφασιστική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση και ένταξη των περιοχών της υπαίθρου ή των καθυστερημένων περιοχών. Θα αναφέρω κάποια αριθμητικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ απλότα. Ο τουρισμός δημιουργεί το 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ποσοστό που φτάνει στο 10% αν λάβουμε υπόψη μας ε, και ε, τις γύρω-γύρω επιχειρήσεις. Είναι περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 10 εκατομμύρια άτομα. 5,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ένωσης και που φτάνει στο 12% αν προσθέσουμε και τις γύρω-γύρω επιχειρήσεις από τον τουρισμό, όχι τις αμυγός τουριστικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο σημαντική τουριστική επιχείρηση, ε, αγορά μάλλον, ε, του κόσμου με 380 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. 42% όλων των αφήξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη είναι μια θαυμάσια πηγή τουρισμών, τουριστών. Ε, η Eurostat είπε το 2008 τα ταξίδια που έκαναν οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε και ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ανεξάρτητα από τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι ένα δικαίωμα το να ταξιδεύουμε σήμερα και να κάνουμε τουρισμό. Και οι διακοπές μας δείχνουν και την ποιότητα της ζωής μας. Δεδομένου της γύρασης του πληθυσμού, θα πρέπει οι τουριστικέ μας δυνατότητε να γίνουν προσπελάσιμες και σε όσου έχουν κινητικά προβλήματα, Παραδείγματο χάρη στους ηλικιωμένου, ε, και σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Οι tour operator ξέρουν ότι αυτό είναι μια πρόκληση. Ε, για το πώς θα εξασφαλίσουν τη μετακίνηση και τις διακοπές σε δεκάδες εκατομμύρια άτομα που έχουν μειωμένη κινητικότητα. Το ίδιο και για τους νέους και για τις διάφορες οικογένειες που έχουν ε, δυσκολίες να επωφεληθούν από τον τουρισμό. Χάρη στην πολιτική μεταφορών και στην υποστήριξή σας ε, προωθώ τα δικαιώματα των επιβατών και ταξιδιωτών. Το δικαίωμα σε όλους να είναι τουρίστες. Και αυτό θα το κάνω με τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας. Ο τουρισμός, όπως και άλλοι του ε, τομείς, επλήγει από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Γι' αυτό το λόγο, κατόπιν τίματός μου, στις 14 και 15 Απριλίου κάναμε μια διάσκεψη στη Μαδρίτη υψηλού επίπεδου για τις προοπτικές ανάπτυξης και επανακίνησης, επανακίνησης του τομέα του τουρισμού ε, υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας. Επίσης έγινε και μια υπουργική άτυπη ε, συνεδρίαση που κατέληξε σε μια κοινή δήλωση των Υπουργών Τουρισμού. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που απέστειλε την κυρία Αγιάλα Σέντερ που μίλησε εξ ονόματος της Επιτροπής και του Προέδρου και συνεισέφερε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες των κρατών μελών. Α πάμε στην κοινή δήλωση, η οποία, την οποία προσυπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων στο τέλος της άτυπης υπουργικής ε, συνάντησης. Ε, καλείται η Κομισιόν στο κείμενο της δήλωσης να υποβάλει μία ανακοίνωση που θα αποτελέσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ε, πολιτική του τουρισμού. Τα κράτη-μέλη δεσμεύονται με τη σειρά τους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς πρόκειται για ένα πρώτο βήμα για την ε, δημιουργία μιας στάσεις που δεσμεύει τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, βιώσιμου, μοντέρνου και κοινωνικά υπεύθυνου. Οι συζητήσεις μας δώσαν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους διάφορους φορείς, ε, δημόσιους και ιδιωτικούς του τομέα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις δικές τους ιδέες για το μέλλον και εκφράζουν τη θέληση να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πολιτική α, τουρισμού. Ε, χάρη σε αυτές τις ιδέες ε, πήρα πολλές ιδέες, ε, έτσι, ιδέες τις οποίες θα ε, διαμορφώσω σε μια πρόταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και που την βοήθησαν να στεφθεί από επιτυχία. Ιδίω θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους βουλευτές που συμμετείχαν στη διάσκεψη, τον κύριο Ρίφ Κράμερ, Λουίς Γκράντες, που δέχτηκαν να μιλήσουν σε αυτή την ε, συνάντηση. Και ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα Σέντερ, η οποία μίλησε μαζί μου στο τέλος ε, και ε, με τον, Υπουργό, τον κύριο Σεμπαστιάν. Λοιπόν, Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θέλω να βάλω στο κείμενο της ε, ανακοίνωσης. Ο βασικός στόχος της πολιτικής τουρισμού θα είναι καταρχήν η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του τουρισμού και η προώθηση της ε, βιώσιμης ανάπτυξής του στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα στόχο που συνάδει απόλυτα με τη νέα στρατηγική Ευρώπη 2020 που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν στις 3 Μαρτίου. Είναι αμφισβήτητο ότι αυτή η ενιαία πολιτική θα ε, εναγκαλίσει όλους τους ενδιαφέρομενους τομείς, την βιομηχανία, την Κομισιόν, ε, που θα συνεργαστούν μεταξύ τους με συντονισμένο τρόπο. Οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις θα είναι συμπληρωματικές των εθνικών μέτρων και θα φέρουν μια προστιθέμενη αξία με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τώρα, για τις διάφορες προτάσεις και σχόλια που ακούστηκαν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, θα προωθήσω ευρωπαϊκές δράσεις γύρω από τους τέσσερις κάτωθι βασικούς άξονες. Πρώτον, να ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του τομέα του τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, προώθηση ενός τουρισμού βιώσιμου και υπεύθυνου στην Ένωση, ε, ειδικά στις αναπτυσσόμενες και αναβιώμενες χώρες. Ενδυνάμωση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προορισμός ποιότητας τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και για τους πολίτες των τρίτων χωρών. Ε, ένταξη του τουρισμού στις πολιτικές και στα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Ένωσης είναι σημαντική για την πρόθεση του τομέα για να αναπτυχθεί δυναμικά και βιώσιμα. Γι' αυτό, κατά την απόψή μου, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις ε, κοινωνικονομικές γνώσεις του τουρισμού και τις συναφείς δραστηριότητε μέσω μελετών, στατιστικών μελετών που θα πρέπει να γίνουν σε στενή συνεργασία με διεθνείς φορείς, παραδείγματο χάρη τη Διεθνή Οργάνωση Τουρισμού και την Οργάνωση για τη Συνεργασία και την Οικονομική Ανάπτυξη. ΩΣΑ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προώθηση ε, πανεπιστημίων, ε, παρατηρητηρίων, δικτύων με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τουρισμού. Οι στατιστικές της Eurostat είναι για μας ε, μια πλούσια πηγή δεδομένων. Και χαίρομαι που η Κομισιόν πρόσφατα υιοθέτησε μια πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού για τις στατιστικές για τον τουρισμό και τώρα ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αποφανθούν επί αυτού του κειμένου. Η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι επίσης ε, στοιχείο κλειδί για την ανταγωνιστικότητα οποιοδήποτε τομέα και του τουρισμού προφανώς. Ιδίω οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των ε, επικοινωνιών είναι σημαντικές για να βοηθήσουν τους πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις τουριστικές ε, υπηρεσίες. Επίσης, νέες τεχνολογίες από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κυρίως ε, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ευαισθητοποίηση, εταιρικέ σχέσεις, ε, πρόσβαση στις πιστώσεις και ενεργή συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Είναι προφανό, προφανές ότι ο εκμοντελισμός της τουριστικής δραστηριότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από μια δέσμευση για να αναπτυχθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες ε, στον τομέα για να διευκολυνθεί η κατάρτιση των ε, επαγγελματιών στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να υπάρξει και κινητικότητα διατομιακή. Η εποχιακότητα είναι ένα άλλο πρόβλημα πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να προωθήσουν την επιμήκυνση της high season, τουριστικής high season στην Ευρώπη. Ε, η πρωτοβουλία Καλυψό που πρότεινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια θαυμάσια ιδέα και την ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υπάρξουν ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών όταν δεν βρισκόμαστε πλέον στη high season. Επίσης, η ποιότητα των τουριστικών προορισμών εξαρτάται από το περιβάλλον και από τις τοπικές κοινωνίες και κοινότητες. Γι' αυτό προτείνω μια σφαιρική προσέγγιση που θα εξασφαλίζει η οικονομική ευημερία, κοινωνική συνοχή, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του πολιτισμού και των τουριστικών ευρωπαϊκών προορισμών. Το νέο ενιαίο πολιτικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίσει και να εξασφαλίσει το σεβασμό των πέντε πυλώνων της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού. Οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική, εδαφική, περιβαλλοντική και πολιτιστική. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να γίνουν θεμελιώδεις και βασικές και πιστεύω ότι πολλοί ευρωπαϊκοί τουρισμοί σέβονται ήδη αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας. Θα ήθελα να αναφέρω Φερρυπίν Κάποιου βασικούς ε, ευρωπαϊκούς ε, προορισμούς που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006. Επίσης, τα δίκτυα τοπικών προορισμών και περιφερειακών προορισμών μέσω της ανταλλαγή ε, καλών πρακτικών και της χρήση δικτών μπορούν να προωθηθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Κομισιόν για να αναπτύξει μαζί με τα ευρωπαϊκά δίκτυα το Next Tour και το δίκτυο των προορισμών ε, μέσω ενός συστήματος δικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να δώσω μεγάλη προσοχή και στην υπεύθυνη συμπεριφορά των Ευρωπαίων τουρισμών απέναντι στο περιβάλλον ε, και στην κουλτούρα, ε, είτε αυτοί είναι τουρίστες στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες δηλαδή, είτε στο εξωτερικό. Ε, εμείς θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα ευρωπαϊκή ποιότητας. Ε, με αυτόν τον τρόπο προωθούμε την ε, εικόνα της Ευρώπης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να έχουμε επαφή με τρίτες χώρες που μπορεί να είναι πηγή τουριστών προς την Ευρώπη και να δώσουμε μια εικόνα της Ευρώπης ως ένα σύνολο τουριστικών προορισμών βιώσιμων και ποιοτικών. Επίσης, η Κομισιό με τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν ε, θα συνεργαστούν επίσης και με, τις εθνικές, με τους εθνικούς φορείς ε, τουρισμού για να αναπτυχθεί από κοινού ένα ευρωπαϊκό σήμα. Αυτό το project έχει την χάνει μεγάλης υποστήριξης και διατράζουν αυτήν την υποστήριξή τους ε, και οι Υπουργοί Τουρισμού που ήταν παρόντες στην άτυπη σύνοδο της Μαδρίτης. Επίσης, η, η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη α, Τουρισμού, το Visit Europe, είναι σημαντική βοήθεια για τους διεθνείς τουρίστες που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη. Πολλές πληροφορίες που αφορούν την Ήπειρό μας και γενικά και τα κράτη-μέλη πιο ειδικά α, δίνονται χάρη σε αυτή τη διακτική πύλη. Επίσης, ε, υπάρχουν και άλλα θεματικά προϊόντα ε, ευρωπαϊκά ευρωπαϊκής διάστασης ή πολυεθνικής διάστασης. Το Visit Europe αφορά τους διεθνείς τουρίστες, τους ξένους τουρίστες. Παρ' όλα αυτά θέλω να προωθήσω και πρωτοβουλίες για να ενδυναμώσουμε την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών προορισμών και απέναντι στους ευρωπαίους τουρίστες. Θέλω να υπενθυμίσω την πρόθεσή μου να παγιώσουμε την συνεργασία στον τουριστικό τομέα με τρίτες χώρες, ε, Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, οι χώρες Κίν, Euromed καθώς και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακριβώς γι' αυτό η Κίνα και η Ρωσία έδειξαν ενδιαφέρον για να ξεκινήσουμε και να ενδυναμώσουμε την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς ε, που συνδέονται με τον τουρισμό. Ιδίω με την Κίνα έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιες πρωτοβουλίες πολύ συγκεκριμένες. Πολύ σύντομα θα υπάρχει μια ε, σύνδεση αμοιβαία μέσω ίντερνετ με την Κίνα ε, για θέματα τουρισμού, ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, σε περιφερειακό επίπεδο για τον βιώσιμο τουρισμό. Αυτό είναι μια ευκαιρία επίσης. Επίσης, στην έκθεση της Σανγκάης θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει την 1η Ιουλίου τα προγράμματά της. Με τη Ρωσία έχουμε έρθει σε επαφή με την Ρωσική Ακαδημία Τουρισμού για να ξεκινήσουμε διάφορες μορφές ε, συνεργασίας. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε την βιομηχανική αρχαιολογία που δίνει τεράστιες ε, δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού. Στην πέμπτη έκδοση της ΕΝΤΕΝ 2010-2011 αναγνωρίζεται αυτό. διάφορα παλιά βιομηχανικά, έτσι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν ε, μεταμορφωθεί, μετασκευαστεί σε, τουριστικές, σε τουριστικούς πόλους έλξης. Θέλω να τονίσω τη σημασία ε, αυτού του, αυτής προσπάθειας. Είναι, είναι καλό οι νέοι μας που σήμερα ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο, με τη μοτοσυκλέτα και έχουν ε, και ένα-δύο κινητά και παρά τις δυσκολίες ζουν σε συνθήκες καλύτερες από τους προγόνους τους, πρέπει να τους πούμε ότι αυτό που έχουν το οφείλουν σε, στις θυσίες χιλιάδων και εκατομμυρίων ε, εργαζομένων Ευρωπαίων που συχνά ε, μετανάστευσαν ε, σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να δουλέψουν στα ορχεία, για να δουλέψουν στα, σε εργοστάσια. Χάρη σε αυτές τις θυσίες η Ευρώπη μας σήμερα είναι μια περιοχή που παρά την κρίση ζει σε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καλύτερες. Και αυτό το οφείλουμε ε, στις θυσίε των προγόνων μας. Ε, αυτό λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα βιομηχανικού τουρισμού θα πρέπει να, να τύχει υποστήριξη. Να μην ξεχάσουμε τις, ε, την ιστορία μας, τις θυσίες των πατέρων μας και να τα γνωρίσουν όλα αυτά τα παιδιά μας. Ο τουρισμός είναι περίπλοκος, ε, οριζόντιος τομέας που χαρακτηρίζεται από οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία που συνδέονται με πολλές ε, πολιτικές. Εσωτερική αγορά, ε, ενεργεία, ε, μεταφορές, κατάρτιση, εκπαίδευση, κουλτούρα, έρευνα, κοινωνία της πληροφορίας, δικαιοσύνη, εμπόριο, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, ανάπτυξη, η γεωργία, εξωτερικές σχέσεις και ανταγωνισμός. Όλες αυτές είναι πολιτικές που συνδέονται με κάποιον τρόπο με τον τουρισμό. Επομένως, θα πρέπει οι υπηρεσίες μου να μην φυστούν κόπον, ούτω ώστε τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού τουρισμού να ενσωματωθούν και στις άλλες κοινοτικέ πολιτικές, προκειμένου οι διάφοροι φορεί του τουρισμού να ενημερώνονται σωστά για τα οικονομικά μέσα που, έχει, που τους προσφέρει η Ένωση, παραδείγματος χάρη το Ταμείο για την Ανάπτυξη Πέθρου, τα διευθυντικά ταμεία, τα ταμεία για τον πολιτισμό, τα ταμεία για την κατάρτιση κτλ. Επίσης θα υπάρξουν συγκεκριμένες γραμμές προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση ε, δράσεων ε, υποστήριξης και συντονισμού ε, για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Θα ήθελα να σε εξασφαλίσω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ενδυναμώσουμε τον τουρισμό στα πλαίσια του προγράμματος για την ε, επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ελπίζουμε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο εργαλείο μέσου ε, για τον τουρισμό στο νέο πολιετές ε, πλαίσιο 2014-2020. Θα ήθελα να σταματήσω μια στιγμή στη δράση που πρόθυσα και προωθώ ακόμα ε, επευκαιρία των ε, προβλημάτων που αντιμετώπισε ο τουρισμός λόγω της ε, κρίσης του Ισλανδικού ηφαιστείου. Στις 15 Απριλίου, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, υπάρχει μια ομάδα εργασίας υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Κάλλας. Οι υπηρεσίε μου επίσης δραστηριοποιήθηκαν για να κάνουμε πρώτη εκτίμηση των ζημιών του τουρισμού. Επίσης, την ε, περασμένη Τετάρτη έκανα μια βιντεοδιάσκεψη όπου συμμετείχαν και οι 27 Υπουργοί Τουρισμού για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και να καθορίσουμε ενδεχομένως ε, κάποιες απαντήσεις συντονισμένες. Από τη συνάντηση που είχαμε τους ε, Υπουργούς προέκυψε μια ανάγκη να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την ανταλλαγή δεδομένων και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον τομέα του τουρισμού στον οποίο θα μπορούσαμε να μπορούσαμε να προσφύγουμε σε περίπτωση που υπάρξουν στο μέλλον νέα προβλήματα λόγω περιβάλλοντος, λόγω μεταφορών ε, ή, λόγω, κάποια πολιτιστικά θέματα. Πολλοί υπουργοί ε, μίλησαν και μου έδωσαν αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε κάποια ε, προκαταρτικά δεδομένα που μου έδωσαν τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η Γαλλία με 260 εκατομμύρια Ιταλία, Ισπανία 200, ε, Ελλάδα 60 είναι οι χώρες που επλήγησαν από την ε, κρίση του ηφαιστείου. Ε, ο τομέας έχασε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ λόγω της κρίσης του ηφαιστείου. Ε, ζήτησα από το ΣΥΜ Κάλλας ε, να συμπεριλάβει το tour operator και τα πρακτορία σε οποιαδήποτε ανακοίνωση θα εκπονήσει η Κομισιόν για το θέμα της ε, κρίσης του ηφαιστείου. Ξέρουμε ότι πέρα από τις αεροπορικές εταιρείες αυτή η άνευ προηγουμένου κρίση είχε άμεση επίπτωση στην, ε, στον τουρισμό. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα έγινε και μία ε, συνέντευξη τύπου για να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι, ηρεμίας και αισιοδοξία, ούτω ώστε ε, να αποκατασταθεί, αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η τουριστική ε, δραστηριότητα. Και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η κρίση λόγω των, του προβλήματος των ε, αεριομεταφορών. μεταφορών. Τώρα, στις 27 ε, Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για ε, τις θρησκευτικές και πολιτιστικές διαδρομές. Η ανακοίνωση για τον τουρισμό 18-19 ε, το Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Τουρισμού στη Μάλτα. Ζητώ συγγνώμη αν φλιάρισα ε, σε αυτή την πρώτη μου παρέμβαση. Αλλά η διάρκεια της παρέμβασής μου ε, είναι ευθέως ανάλογη με τη σημασία του τουρισμού. Είναι ένας οικονομικός τομέας που δεν είναι σε καμία περίπτωση δευτερεύον. που δεν είναι δευτερεύον ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου έδωσε ο πρόεδρος Μπαρόζο, αλλά πολύ σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για αυτή τη δήλωση. Ιδιαίτερα το κομμάτι που φορούσε τη βιομηχανική κληρονομιά. Έχω ένα μεγάλο κατάλογο ομιλητών, 15 προς το παρόν, οπότε κατανοείται ότι θα πέσει ράβδος κατά του, της συζήτησης αυτής. Προτείνω λοιπόν τρία λεπτά για τους εκπροσώπους των ομάδων και δύο λεπτά για τους βουλευτές τους υπόλοιπους. Σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτό το χρόνο και θα κάνουμε γύρους απαντήσεων μέχρι 7 ερωτήσεις. Αντί να απαντήσει όλες τις 15 ερωτήσεις ο, ο, ο Επίτροπος. Και ξεκινάμε με τον κύριο Πασκουάλ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ταγιάννη, καλώς ορίσατε στο σπίτι σας. ότι είναι ένα γεγονό που διατηρείτε αρμοδιότητε που σα επιτρέπουν να επιστρέψετε στο σπίτι σα. Βλέπω όμω ότι αυτέ οι αρμοδιότητε μετατίθεται πια από το θεωρητικό επίπεδο στο πρακτικό μέσω τη νομική βάση. Και είναι ότι αυτή η νομική βάση, συγκεκριμένα το 195 άρθρο, είναι πολύ περιοριστικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε αυτές οι αρχές αναλογικότητας και της επικουρικότητας που απαιτεί η συνθήκη να τηρούνται και να μην προκαλούνται προβλήματα και ζήλιες μεταξύ των χωρών μελών σοφράς αρμοδιότητες. Είναι λοιπόν ε, ευτυχές το γεγονός ότι ασχολείστε εσείς με αυτό το γεγονός γιατί για μια φιλόδοξη πολιτική τουρισμού θα χρειαστεί πολλή διάλογο και μεγάλη συνένεση μεταξύ όλων των χωρών μελών, ώστε να μην υπάρχει καμία παρέμβαση όσον αφορά τις ίδιες αρμοδιότητες και ξέρουμε ότι πολλές φορές αυτοί οι δισταγμοί οδηγούν στο ότι οι χώρες που ασχολούνται με τον τουρισμό βλέπουν στους υπόλοιπου ανταγωνιστές. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο, έστω και είμαστε ανταγωνιστές, να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκές τουριστικές πολιτικές που θα είναι θετικές. Ο χρόνος μου έδωσε ο πρόεδρος Σίμψον ελάχιστος, γι' αυτό δεν θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα, τα σημαντικά που θα ήθελα να δείξω. Αυτή είναι η να κάνουμε. Πάντως όλα αυτά που είπατε τα προσπογράφω από το α μέχρι το ω. Νομίζω ότι αυτά που είπατε ήταν ευφυή, ήταν προσεκτικά, αλλά ήταν και ταυτόχρονα φιλόδοξα. Πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν, χωρί βεβαίω να παρενεύουμε, όπω έλεγα προηγουμένω, στι ίδιε τι αρμοδιότητε των χωρών μελών. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το θέμα αρμοδιοτήτων που μας παρέχει η συνθήκη είναι πιθανό να υποστηρίξουμε, να συντονίσουμε, να συμπληρώσουμε τα μέτρα από τις χώρες μέλη μέσω πρωτοβουλειών πολυεθνικής ή πανευρωπαϊκής διάστασης και στη συνεργασία με τοπικές επίση ε, πρωτοβουλίε. Αυτά τα λέω εγώ. Τα λέει η ίδια η Κομισιόν που στην ανακοίνωσή της για την έξοδο ε, διαβουλεύσεων ήταν αρκετά συνετή στην περιγραφή ακριβώς του πεδίου της αποστολής της. Και εσείς πολύ σωστά καταστήσατε σαφές πώς αυτή η στόχη για την ανάπτυξη του τουρισμού, για την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας, για την πρόθεση της Ευρώπης σε άλλες αγορές, όλα αυτή η στόχη λοιπόν θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτευχθούν στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων. Εγώ, απλά και μόνο, να πω ότι είναι θετικά τα εργαλεία που έχουμε, να αναφέρω και κάποια που είναι σημαντικά για την Ισπανία, αλλά και για άλλες χώρες όπως η Ιταλία και άλλες χώρες που θα ήθελαν να έχουν παρόμοιες εμπειρίες ή καλυψώ ας πούμε ως μια πολιτική δηλαδή ολοκλήρωσης και ένταξης της τρίτη ηλικία, κάτι το οποίο θα ανοίξει ένα πεδίο το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήταν καλό να φανταστούμε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα μπορούσε να, να συνδυάσει την προώθηση τη Μάρκα Ευρώπη χωρί ανταγωνισμό μεταξύ των άλλων εμπορικών σημάτων. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να εξετάσουμε νέου προορισμού, τουριστικού, Το πεδίο είναι πολύ φιλόδοξο, εσείς το περιγράψατε με πολύ σαφή λόγια. Εγώ το προσυπογράφω και επειδή κύριε Σίμψον μου τελειώνει και χρόνο, να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη για τα λόγια του και έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε και να εργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αλχαντραουή, τρία λεπτά για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για αυτά τα οποία μας είπατε. Πράγματι ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός τομέας, οπότε και οι μεταφορές ε, έχει, έχουν μεγάλη επίπτωση στον ε, τουρισμό και με την έκρηξη, είδα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος για να μπορέσει να βρει μια εναλλακτική λύση μετακίνησης, τα δικαιώματα των επιβατών ε, και το πώς θα αντιδράσουν ε, τυχόν συλλογικά. Οπότε είδαμε επιπτώσεις που πάνε και πέρα από τον τουρισμό σημείωσα αυτό το οποίο είπατε για ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αηφορίας του τομέα, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε συγκεκριμένα να δούμε τι περιμένουν από μας οι άνθρωποι και εγώ ε, θεωρώ πως υπάρχουν κάποια πράγματα που εντάξει μπορεί να είναι λίγο εκτός των αρμοδιοτήτων τας, αλλά θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για τον ε, σιδηρόδρομο, για όλα τα μέσα μεταφοράς. Επίσης η ευκολία διάδοση των πληροφοριών που σχετίζεται με αυτό. Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν οι καταναλωτές. Ε, Παραδείγματο χάρη η εναρμόνιση των κριτηρίων για τα αστέρια των ε, ξενοδοχείων. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και αντιλαμβάνομαι πως βέβαια στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θίξατε είναι η αποτελεσματική χρήση των ε, δυνατοτήτων ε, στη high season και τη low season και πρέπει εδώ πέρα να το δούμε αυτό και να συνδεθεί αυτό βέβαια οπωσδήποτε και με τη γύρανση του πληθυσμού καθώς πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτοι στις περιόδους στις οποίες θα πάνε διακοπές. Τέλος, αυτό το οποίο είπατε, η μάρκα Ευρώπη, το σήμα Ευρώπη και τη σχετική πύλη πρέπει να είναι πράγματι σαφές ε, να υπάρχει εκεί πέρα ένα κομμάτι πόλης, ένα κομμάτι πράσινος τουρισμός, ένα κομμάτι βεβαίως για τις ε, παραλίες κτλ. Τέλος έχω την αίσθηση πως πράγματι θέλετε να επιτύχετε κάποια πράγματα και θα φτάσετε λίγο έτσι στα όρια εάν θέλετε της αρχής της επικουρικότητας. Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει κάποια εναρμόνιση για να δοθεί μια όθηση στον ε, τουρισμό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτά τα οποία μας είπατε. Με πρόλαβε σε αρκετά σημεία ο κύριος Ελχαντραούι. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό τομέα ο τουρισμό και στην συνθήκη τη Λισαβόνα. Τώρα έχουμε μεγαλύτερε αρμοδιότητε, τι οποίε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Πολλοί δεν ξέρουμε ότι έχουμε αυτέ τι νέε αρμοδιότητε. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία που είναι και ερωτήσεις. Είπατε πως θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκλήρωση πολιτικών και των χρημάτων για τον τουρισμό και εκεί πέρα είπατε πως θέλετε να συνδεθούν τίτλοι του υπερβολισμού που σχετίζονται με τον τουρισμό. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα, καλό θα ήταν αυτό, αλλά τι αναμένετε από πλευράς ε, χρηματοδότησης, ε, τι είναι δυνατόν, έχετε συγκεκριμένα νούμερα κατά νου ή θα ζητήσετε περισσότερα λεφτά για τον τουρισμό. Δεύτερον, ε, αναφέρατε την ε, πληροφορική, ναι πράγματι εκεί πέρα είναι σαφής η σύνδεση με τις ε, μεταφορές ε, και γι' αυτό το βρίσκω κρίμα πως έχουν διαχωριστεί αυτά τα πράγματα εντός της Κομισιόν. Θα πρέπει νομίζω ο τουρισμός να παραμείνει στις μεταφορές γιατί είδαμε και με τη στάχτη πως τα δικαιώματα των επιβατών σχετίζονται άμεσα με την πληροφορική και με τη γενικότερη πληροφόρηση όπως είπε ο κύριος Ελχαντραουή και με τα τρένα και με τις αναλλακτικές είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε ε, στον σημερινό τουρισμό να μπορεί ο καθένας να κινηθεί δηλαδή ανεξάρτητα έχοντας ε, ε, μια καλύτερη εικόνα από το ίντερνετ. Τώρα είπατε πως θέλετε να επιμικίνετε την high season. Αυτό γίνεται ε, μέσω της κλιματικής αλλαγής, όπως άλλωστε γίνεται πιο μικρή η περίοδος του χιονιού και και με το σύστημα αυτό καλύψω πώς συνδέεται. Επίσης μιλήσατε για την ε, αηφορία. Νομίζω πως εδώ πέρα θα πρέπει να ζητήσετε και από τα κράτη-μέλη να δώσουν μεγαλύτερο βάρος όταν μιλάμε δηλαδή για ευρωπαϊκό τουρισμό, για ανάπτυξη μιας αγοράς και μια πολιτική μεταφοράς προς νέες αυτές αναψώμενες χώρες. Μιλήστε επίσης για τις 27 Σεπτεμβρίου για μια ημέρα ταξιδιού πολιτισμικού και θρησκευτικού. Τι ακριβώς ε, σημαίνει αυτό και τι ακριβώς αναμένεται. Σας ευχαριστώ για την πράσινους ο κύριος Κράμερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ για αυτά που μας είπατε. Αναφέρατε πολλές φορές πως είναι σημαντική η αηφορία και πρέπει να αποφευχθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα επιμείνω κι εγώ. Ο τουρισμός του αύριο είτε θα είναι αηφόρος είτε δεν θα υπάρχει. Έχουμε ακτές ε, στη Μεσόγειο που καταστρέφονται από τον τουρισμό. Το αναφέρατε και αυτό και δεν πρέπει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ο φόρος τουρισμός είναι σημαντικός γιατί και ο στόχος ε, της Ένωσης είναι να μειωθούν οι εκπομπές. Πώς συνεργάζεστε εδώ πέρα με τους άλλους επιτρόπους, τι θα συνεισφέρει συγκεκριμένα ο τουρισμός για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αναφέρατε τα δικαιώματα των επιβατών Έχουμε το μειονέκτημα εδώ πέρα πως ε, δεν μπορεί κανείς να βάλει στα γρήγορα τρένα το ποδήλατο. Εδώ και χρόνια, δεκαετίες, ε, ανθεί ο ποδηλατικός τουρισμός, αλλά μάλλον δεν το έχουν καταλάβει αυτό οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι. Τι κάνετε για να το εφαρμόσετε αυτό στην πραγματικότητα, ότι θα μπορεί κανείς να πάρει το ποδήλατό του σε όλα τα τρένα. Αναφέρατε επίσης την ιστορική αρχαιολογία, Αυτά τα οποία αναφέρατε με τα ορυχεία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα τα βλέπουν αυτά οι επόμενες γενιές και ενδιαφέρον είναι να βλέπουν και το σίδηρο παραπέτασμα. Ξέρετε πως υπάρχει το μονοπάτι εκεί πέρα του παραπετάσματος όπως λέγεται το οποίο εγκρίθηκε από, την, ε, εγκρίθηκε από μας πρόσφατα. Θα φροντίσει να το αυτό και η Κομισιόν και το Συμβούλιο επίσης να φροντίσει έτσι ώστε οι ποδηλατόδρομοι, τα 17.000 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων που υπάρχουν ε, στην Ευρώπη να ενσωματωθούν στα δίκτυα μεταφορών καθώς ε, αυτό προσφέρει πάρα πολλές ε, ευκαιρίες ε, και στις χώρες αυτές του πρώην παραπετάσματος. Ήμουν δε πρόσφατα στην ε, Μακεδονία που υπέγραψε ένα μνημόνιο με την Βουλγαρία ακριβώς για αυτές τις πάρα πολύ απομακρυσμένες περιοχές και θέλω να τους προσελκύσουν με την ιστορία Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση με τους ε, άλλους επιτρόπους, γιατί εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολλές ε, αρμοδιότητες ε, οι οποίες είναι κοινέ και αυτό αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση. Π.χ. στον τομέα της κοινωνίας 60% πηγαίνει στην οδοποιία αλλά αν το επικεντρώσουμε νομίζω στον αηφόρο τουρισμό θα υποφεληθείτε και εσείς πολύ περισσότερο ως Επίτροπος ε, Τουρισμού. Ευχαριστώ κύριος Κάντσιαν. Τελευταίος για δύο λεπτά. Δύο λεπτά κύριε Κάντσιαν. Sorry. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που είναι εδώ ο συνάδελφος Ταγιάννη και το απευθύνω τις ευχές μου για καλή δουλειά σε αυτό το νέο θέμα που νομίζω ότι πολύ σωστά έχει ενταχθεί ως τρίτη οικονομική δύναμη στις ε, ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Μίλησε για αυτή την οικονομική, μάλλον για αυτή την ευρωπαϊκή ανάπτυξη πρέπει να είναι ευφυής, βιώσιμη και διατηρήσιμη. Νομίζω ότι πολύ σωστά λοιπόν έδωσε έμφαση σε αυτούς τους τρεις πυλώνες ε, ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουρισμού. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να επιμείνω πάνω σε αυτό είναι ότι με τη σωστή συμπληρωματικότητα και τη σωστή επικουρικότητα με τις εθνικές ε, ε, με τις χώρες μέλη που ανέφερε και ο κύριος Σταγιάννη είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου η υπηρεσία που παρέχεται στον ε, τουρίστα να είναι κατά κάποιο τρόπο κατανεμημένη. Και αναφέρομαι βεβαίως εδώ στις διαδρομές και αναφέρομαι εδώ στις ε, διασυνδέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανά περιοχή και ένα είδος περιοχής. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ο κ. Σταγιάννη στις διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις οδούς δηλαδή στις μεγάλες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εγώ επ' αυτού θα ήθελα να δαπανίσω περισσότερο χρόνο και διαθεσιμότητα. Και το δεύτερο αίτημα που έχω είναι η απλούστευση και η τρίτη είναι η συμπλήρωση η ολοκλήρωση μόνο των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών που έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας και άλλη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, θέλετε να ξεκινήσετε με αυτά τα προδόρπια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επίτροπος του τουρισμού από τι 9 του Φλεβάρι. Δεν γίνεται σε λίγους μήνες να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω κάποια προγράμματα και να σας πω κάποια πράγματα για το τι έχω κάνει δηλαδή σε αυτή την σύντομη χρονική περίοδο που έχω αναλάβει. Να ξεκινήσουμε κάποια σημεία αρχών. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στην επικουρικότητα και στην ε, σχέση της προώθησης του τουριστικού προϊόντος σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό εξάλλου συζητήθηκε και στην άτυπη συνάντηση υπουργών στη Μαδρίτη και επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν έχω πουδενή πρόθεση να παρισφρήσω ή να καπελώσω τις αρμοδιότητες των χωρομελών ή να τις μειώσω. Αντίθετα, θέλω να προσπαθήσω και να κάνω προσπάθειες ώστε οι πολιτικές κομισιόν αποτελεί μια προστεθέμενη αξία στις πολιτικές των χωρομελών, δηλαδή να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να έχουν το κάτι παραπάνω. Είχαμε μια συμφωνία που υπέγραψε η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία για συνεργασία στον τουριστικό τομέα. Και οι τρει υπουργοί που συνάντησα ξεχωριστά και δημερό στη Μαδρίτη όλοι, όλοι ζητούσαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδεχομένω για να επεκταθεί και η συμφωνία αυτή και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δηλαδή είδα ιδιαίτερη ευαισθησία α πούμε από την ε, Βελγίδα Υπουργό Τουρισμού και ενδιαφέρον για αυτή τη συμφωνία. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή συνεργασία για τον τουρισμό σημαίνει ότι υπάρχουν 10 ας πούμε τουρίστε που πάνε στην Ισπανία, 10 που πάνε στη Γαλλία, 10 που πάνε στην Ιταλία και με τη βοήθεια τη Ευρώπη θα μπορούσαμε να προσθέσουμε άλλου 10. Δηλαδή, τρει φορέ το 10 δεν είναι 30, αλλά 40. Και αυτό σα το δίνω έτσι ω απλοϊκό παράδειγμα του δικού μου του στόχου. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε και ε, εκδηλώσεις όπως είπα κατά τη διάρκεια της ακρόασης και εκδηλώσεις που γίνονται παγκοσμίω, αλλά και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολυμπιακή Λονδίνου, ε, έκθεση Μιλάνου 2015. Δηλαδή να κάνουμε προσπάθειες ώστε αυτές οι εκδηλώσεις να αποτελούσουν ένα είδος όθησης για την αύξηση του αριθμού των τουριστών στις, στο Λονδίνο θα έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχουμε εκατομμύρια άτομα τα οποία θα φτάσουν εκεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες οπότε γιατί να μην προσπαθήσουμε λοιπόν να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών στο Λονδίνο προβλέποντας, ας πούμε τη χρήση του αεροπλάνου ή του σιδηροδρόμου για επισκέψεις στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Για την έκθεση του Μιλάνου, γιατί να μην αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών που θα έρθουν ας πούμε από την Άπα Ανατολή μέσω προγραμμάτων που βεβαίως εκτός από την ε, πτυχή της ε, εργασίας, δηλαδή να προσπαθήσουμε να γίνουν επισκέψει από το Μιλάνο στην Τεριά, Τεριά, στη Βενετία, Βενετία, Βουδαπέστη. Δηλαδή να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η Ευρώπη να αποτελεί μια προστιθέμενη αξία. Εγώ που δεν θέλω να παρανεύω στι ε, εθνικέ πολιτικέ στο χώρο μέλλον. Θέλω απλά και μόνο το ξαναλέω αυτό το 3 φορέ 10 αντί για 30 να κάνει 40. Ώστε η Ευρώπη τέλο πάντων ώστε να είναι αυτή η προσθέμενη αξία και να εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς. Δεν θέλω λοιπόν ε, που δεν είναι να παραβιάσω τις αρχές της πικορικότητας και θα ήθελα να πω ότι ήδη στην δεύτερη συνάντηση είδα μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον από τους υπουργούς τουρισμού που είδαν και εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Ένωση και εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους υποστηρίξει. Όχι να παρενέβει, να παρισφρήσει, να καπελώσει τις αρμοδιότητες τους, αλλά να αξιοποιήσει και να αξιολογήσει την εργασία τους. Αυτό θα ήθελα λοιπόν να είναι το έργο μας. για να βρούμε και συμφωνίες. Εγώ δεν θα ήθελα να επιβάλλω κάποια έτσι ολοκληρωμένα ή κοινά εισιτήρια ή τέλο πάντων να εναρμονίσω τον ουρανό και τα άστρα. Απλά και μόνο θέλω να βρω συμφωνίες μεταξύ χωρομελών που να ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ό,τι θα κάνω εγώ θα αποβλέπει στην ανέβρεση συμφωνιών μεταξύ των χωρομελών που θα αξιοποιεί την κληρονομιά της κάθε χώρας. Ό,τι μπορώ θα το κάνω. Επί παραδείγματι στην ανακοίνωση που προετοίμασα ως Επίτροπος Τουρισμού για τις αστικές μετακινήσεις υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία εκεί και εγώ είμαι πεπισμένος ότι η σχέση μεταξύ τουρισμού και μεταφορών είναι ουσιώδης. Και μάλιστα ακούσαμε και κάτι για τα δικαιώματα των επιβατών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και μάλιστα αν αυτοί μετατρέπονται και σε τουριστές αυτό νομίζω είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και αυτό δεν αφορά τι δικέ μου μόνο αρμοδιότητε ω επίτροπο, αλλά από πρακτική σκοπιά το γεγονό ότι ήμουν βεβαίω και επίτροπο μεταφορών θα διευκολύνει και τη δουλειά μου ω επίτροπο τουρισμού και όπως ήδη έχω πετύχει σημαντικά αποτελέσματα για ε, τους ε, Ευρωπαίους πολίτες νομίζω ότι τα ίδια θα κάνουμε και στο, στο νέο αυτό πεδίο αρμοδιοτήτων μου. Όσον αφορά το άλλο θέμα που έθεσα στην προσοχή σας και που ο κύριος μέσνερ έθιξε. Κάποτε λέγανε ότι, ότι το χρήμα κάνει τον πόλεμο, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι το χρήμα κάνει και τον τουρισμό για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας και στην ε, ομιλία μου μίλησα για την εδραίωση κάποιων γραμμών του προπολογισμού που αυτή τη στιγμή αφορούν χωριστά κάποιες δράσεις υποστήριξης και για συντονισμό των πολιτικών. Θα έπρεπε λοιπόν να διασφαλίσουμε μια συγκεκριμένη ενίσχυση του τουρισμού μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας τη Κομισιόν και εδώ ακριβώ ζητώ την ε, δική σα υποστήριξη και του Συμβουλίου ώστε να περιλάβουμε και ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τον ε, τουρισμό στο πολιετε πλαισιο πλαίσιο 2015-2020. Θα μπορούσαμε λοιπόν από κοινού να εντοπίσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτές είναι οι ιδέες μου. Βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μετά τη δουλειά τους επόμενου και για την ανακοίνωση για τον τουρισμό και θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να βρω κάποια σαφή στοιχεία ακόμα σε συνεργασία με τις χώρες μέλη αλλά και με εσά. Οπότε οποιαδήποτε δική σας ένδειξη, πρόταση, συμβολή πέραν αυτών που έδωσε η Κομισιόν γενικότερα για μέ θα είναι ε, πολύτιμη. Όσον αφορά και την ολοκληρωμένη προσέγγιση εγώ θα προσπαθήσω να μελετήσω όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρξουν λύσεις τις οποίες θα συμμερίζονται και οι συναδελφοί μου επιτροπή σε άλλους συναφείς τουρισμούς. Όσον αφορά τώρα τον βιώσιμο τουρισμό, εγώ στην ομιλία μου μίλησα για δείκτες βιωσιμότητας. Θα μπορούσαμε παραδείγματι να προβλέψουμε μια μπλε σημαία όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που έχουν ιδιαίτερη αξία όσον αφορά την περιβαλλοντική σκοπιά. Αυτό είναι μια ιδέα. Βεβαίω όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε ανάπτυξη του τουρισμού αν συνεχίσουμε να καταστρέφουμε το, την περιβαλλοντική μας κληρονομιά. Γιατί η κερδοσκοπική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος μπορεί ενδεχομένω να δίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα πλούτη σε κάποιους, όμως μακροπρόθεσμα βλάπτει την οικονομία. Οπότε θα πρέπει και αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη. Και κάποια άλλα πράγματα που υπόθηκαν να σχολιάσω, ο κύριος ε, Κράμερ γνωρίζει ότι έχω αναλάβει σοβαρέ δεσμεύσει για τα δικαιώματα των ε, ποδηλάτων και ως Ευρωπαίος Επίτροπος θα συνεχίσω να εργάζομαι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη του τουρισμού με το ποδήλατο, που είναι ένα από τομεί που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη και το γνωρίζω άμεσα αυτό, γιατί στην χώρα μου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού. Θα πρέπει να προβλέπουμε βεβαίω κάτι και για τα θέματα των μεταφορών αλλά βεβαίως νομίζω ότι χιλιόμετρα ας πούμε ποδατοδρόμων αποτελούν πράγματι μια σημαντική αξία, πολιστική αξία για την Ευρώπη. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιε απαντήσει. Ε, Βεβαίω στη συνέχεια είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να μαθήνουμε σε όλα τα θέματα τα οποία α, θίξατε σήμερα στη συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να λάβω ενδείξει από εσά αν θέλετε να τι υποβάλλετε γραπτώ ή αν θα ήθελε ο πρόεδρο να τις αποστείλει επισήμω ω συμβολή τη Επιτροπή σα στην εργασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή για την Αγγλική Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιο ότι θα το πράξουμε αυτό. Και εγώ ω πρόεδρο τη Επιτροπής χαίρομαι που υπάρχουν έτσι ε, και σύντομε απαντήσει. Πόμε μιλητής, κύριε Σέντερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να συμφωνήσω με τα λόγια του συναδέλφου Λίου Δεγκράντες για την χαρά και την ικανοποίηση που εξέφρασε που είστε εσείς κύριε Ταγιάννη υπεύθυνο και αρμόδιο για την πολιτική τουρισμού. Όπω είπε ο κύριο Μάσνερ, ο τουρισμό δεν έχει διαρρεθεί. Βρισκόταν την ε, Επιτροπή Βιομηχανία, αλλά ήταν ε, το άσχημο παπί της υπόθεσης. Ο κύριος Φερχόγγεν από την αρχή είπε ότι δεν ήταν και τόσο βιομηχανική η πολιτική ευθεία, Αναγνώριζε βέβαια στην αξία τουρισμού, αλλά δεν ήταν τόσο βιομηχανική η πολιτική. Έλειπε βέβαια και νομική βάση, αλλά έλειπε και η πολιτική βούληση, που νομίζω ότι οι υπάλληλοι τη Κομισιόν αναπλήρωσαν εν μέρη με την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, γιατί οι πρωτοβουλίε ΕΔΕΜ και Καλυψό ή για, το, για τον ποδηλατικό τουρισμό, το βιώσιμο, όλα αυτά ακριβώ ήταν τμήμα των πρωτοβουλειών που είχε υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, ώστε ο τουρισμό να μην ε, πεθάνει από αδράνεια. Γι' αυτό ακριβώ είχαμε τύχει να είναι ο κύριος Σταγιάννη που ξέρει πολύ καλά αυτή την Επιτροπή λόγω των προηγούμενων θέσεών του και ασχολείται τώρα με τον τουρισμό με τρόπο έτσι ενεργό. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά η, η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη γιατί θα πρέπει ακριβώ να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη διαφορετικά ενώπιον αναδειωμένων δυνάμεων των τουρισμών που έχουν δυνατότητα marketing πολύ σημαντική σε επίπεδο εμπορικό, σε επίπεδο οικονομικό και βέβαια σε επίπεδο τουριστικό, εκεί ενδεχομένω θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε αδύναμη θέση. Και βεβαίω ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν για ένα πρόγραμμα πολιετές και θα ήθελα να σα ρωτήσω δύο πράγματα σχέση με τι ιδέε που έχετε. Όταν μιλάμε για ποιότητα στον τουρισμό μιλάμε για του ανθρώπινους πόρου, δηλαδή για την επαγγελματικότητα των ανθρωπίνων πόρων, των εργαζομένων δηλαδή, κάτι το οποίο σε κάποιου τομεί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας αφορά μέσα. Να σας ρωτήσω κάτι επίσης, κάτι για την διαφοροποίηση του πλούτου της Ευρώπης σε σχέση με τον τουρισμό. Δηλαδή να κάνουμε επιμέρους τουρισμούς, όπως γαστρομικός τουρισμούς, πέρα δηλαδή από τον πολιτισμό ή άλλες μορφές τουρισμού, να κατεβούμε δηλαδή πιο κάτω σε επίπεδο εξειδίκευση ώστε να αναζητά ένα συγκεκριμένο στοιχείο ο τουρίστας θα κάνει τουρισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Πελπάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε Συμφωνώ με τους ε, στόχους που έχετε θέσει και με τις κατευθυντήρες γραμμές στο πρόγραμμα. Θα ήθελα όμως να σας ε, ρωτήσω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι ο τουρισμός στην Ευρώπη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και καινοτόμος αν μπορούμε να ενσωματώσουμε μια έτσι διαφορετική σκοπιά. Θα ήθελα λοιπόν στα προγράμματά σας, σε όλα τα έγγραφα τα οποία θα εκπονήσετε, να κάνετε μια ιδιαίτερη μνήμα στην ανάγκη προσαρμογής όλων αυτών των πολιτικών για τα άτομα με, με προβλήματα ή με μειωμένη κινητικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένας, ένας ε, δείκτης διαφοροποίησης, γιατί σχετίζεται με αυτό που είπατε προηγουμένως και εσείς για την κοινωνική βιωσιμότητα. Κάνω λοιπόν ένα αίτημα συγκεκριμένο για την ανάπτυξη και αυτού του στοιχείου. Δεύτερο θέμα η επαγγελματικότητα. Νομίζω ότι ο τομέα του, ευρώ, του τουρισμού στην Ευρώπη μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με την κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό όμω απαιτεί προσπάθειε ακριβώ για να αξιοποιηθεί το επάγγελμα του εργαζόμενου στον ε, τουριστικό τομέα και να δίδεται μια συγκεκριμένη κατάρτιση, ενδεχομένω και ακαδημαϊκή, που νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Τρίτον, θα ήθελα σε όλα τα θέματα του τουρισμού να λαμβάνεται υπόψη σε περιφέρειες, να λαμβάνει υπόψη και περιφέρειες οι οποίε έχουν αρμοδιότητε και οι οποίε έχουν αναπτύξει πολιτικέ για τον τουρισμό. Θα πρέπει να σα ρωτήσω επίση κατά πόσο λάβετε υπόψη στο το θέμα τη ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και ξέρω ότι αυτό σχετίζεται με τα ε, θέματα τη γεωργία, αλλά η ανάπτυξη τη υπαίθρου θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι κοινωνική, θα πρέπει να περιλαμβάνει βιωσιμότητα περιβαλλοντική. Με όλε αυτέ τι επιχειρήσει που περιλαμβάνει και που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις ενισχύσεις και τις ε, βοηθήσεις που αναφέρατε κι εσείς. Και να πω ότι συμφωνώ και με την κυρία Αγιάλα ότι είναι απαραίτητο να καθορίσουμε διαφορετικές διαδρομές, επί παραδείγματι αυτές που σχετίζονται ε, με το Νίνο. Γιατί η Ευρώπη νομίζω έχει μεγάλη δυνατότητα δημιουργία δικτύων τα οποία θα είναι πάρα πολύ ελκυστικά, τα οποία παρουσιάζουν νέε δυνατότητε. Ευχαριστώ. λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχει μια νέα τάση περίπου ε, στα επίπεδα, στο επίπεδο του τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός το 1997 δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο ε, για τη συνεργασία του Λουκά του Λουξεμβούργου με το Συμβούλιο της Ευρώπης και δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα με θεματικές διαδρομές το χάρη το προσκύνημα στην Ανδαλουσία ε, το, η διαδρομή για την ελιά, ε, για το μετάξι κτλ. Η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή του Κοινοβουλίου ε, για τη Μεταφορές και τον Τουρισμό πρότεινε μία έκθεση για τον τουρισμό και την εταιρική σχέση για τον τουρισμό στην Ευρώπη ε, για να προωθηθούν διάφορες ε, πρωτοβουλίες για τουριστικές διαδρομές στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Πώς πιστεύετε ότι οι πολιτιστικές διαδρομές, οι ιστορικές διαδρομές και οι θρησκευτικές διαδρομές με, το, με την ετικέτα του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να προωθήσουν μια διασυνοριακή προσφορά τουριστική στην Ευρώπη, θεματικής και μια θεματική διάσταση. Ποια είναι η γνώμη σας για τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα προγράμματα πολιτιστικών διαδρομών για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ορατότητα, για να προωθηθεί ο υπεύθυνο και διοντολογικός τουρισμός, κοινωνικός, ε, περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, καθώς και οικονομικά βιώσιμος. Αυτοί οι τελευταίοι στόχοι ακούστηκαν και στη διάσκεψη, όπως είπατε και εσείς, στις 15 Απριλίου. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Κάποια σχόλια. Καταρχάς, ε, καλή επιτυχία, κύριε Ταγιάννη, γιατί η πρόκληση που αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλη. Ε, το θέμα της επικουρικότητας το ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι. Επιβαρύνται, θα έλεγα, ε, από το γεγονός ότι συχνά οι εθνικές αρμοδιότητες μπλέκονται με τις αρμοδιότητες των περιφερειών και αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο πολύ διαφοροποιημένο, δύσκολα εναρμονίσιμο και επομένως ε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη-μέλη θα αντιμετωπιστούν και από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια... Άκουσα με μεγάλη χαρά την πρόταση για το ευρωπαϊκό σήμα. Καλό είναι να το προωθήσουμε. Θα πρέπει να το οικοδομήσουμε γύρω από μια πραγματική βιώσιμη βιομηχανική πολιτική και νομίζω ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Ε, επίσης, με μεγάλη χαρά άκουσα αυτό που είπατε για τις μεγάλες διεθνείς διασκέψεις, την Expo 2015 και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, η Ολυμπιακή κτλ. Ε, θα μιλήσουμε σε διάφορες ακροάσεις για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διοργανώσεις για την πρόθεση του ευρωπαϊκού τουρισμού. Και ένα ερώτημα. Τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες ε, παρουσιάσετε μια τελευταία ανακοίνωση για το θέμα των καθαρών και αποτελεσματικών σε ενεργειακό επίπεδο οχημάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Εσείς θεωρείτε ότι συνδέεται με την αστική κινητικότητα αυτή η προσπάθεια και με την προσπάθεια ανάπτυξης του αστικού τουρισμού, του τουρισμού δηλαδή της πόλης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαβίσα, δύο λεπτά. Η κυρία, μάλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η έκθεσή σας είχε πάρα πολλές φιλόδοξες ιδέες. Τις άκουσα με χαρά. Θέλω να σας υποβάλω μια ερώτηση. Που είσαστε, ε, σε εσά που είσαστε και πρώην Επίτροπος Μεταφορών. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπατε για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και για ανθρώπους που δεν είναι τόσο πλούσιοι στην Ευρώπη. Και αυτά που είπατε για επενδύσεις σε βιώσιμες και εναλλακτικές σε βιώσιμους και εναλλακτικού τρόπους τουρισμού. Ίσως η ερώτησή μου είναι λίγο αγενής, αλλά θα την κάνω παρόλα αυτά. Για τους ε, πιο φτωχούς ανθρώπους, πώς θα δημιουργήσουμε τις δυνατότητε για να επισκεφτούν, ας πούμε, το μεσαιωνικό Τάλιν. Οι βαλτικές χώρες βρίσκονται ακόμα πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, γιατί δεν υπάρχουν συνδεδομικές μεταφορές που να τις συνδέουν με άλλες χώρες. Πιστεύετε ότι ένας βαλτικός σιδηρόδρομος πρέπει να τύχει υποστήριξη από την Ευρώπη, γιατί αυτό το πρόγραμμα χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης μπορεί να μην τελεσφορήσει. Μπορεί δηλαδή άλλα κράτη-μέλη να μην το υποστηρίξουν. Έχω και άλλους ομιλητές στον κατάλογο και θα τον κλείσω τον κατάλογο. Εγώ θέλω να καταλάβω πόσους έχουμε για να διαρρώσω το χρόνο. Ε, όταν εσείς ε, τελευταία στιγμή ξυπνάτε και ζητάτε να μιλήσετε, ε, μου δημιουργείται πρόβλημα με τον υπολογισμό του χρόνου. Τσικάου, Λιμπεράτσκι, Κουμουτσάκος, Σαββάνα και Κρίσβακ και τέλος και ο Πρόεδρος. Πρώτα θα απαντήσω όμως ο Επίτροπος και μετά θα ακούσω τους υπόλοιπους ομιλητές. Θα απαντήσω και στην Αγία Λασέντερ και στην κυρία Μπιλμπάου και στους τελευταίους ομιλητές. Για, την, για αυτό που η κυρία Αγία Λασέντερ και η κυρία Μπιλμπάου καταρχήν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε διάφορα είδη τουρισμού. Είναι σημαντική, σημαντικός πόρος ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια τεράστια αρχαιολογική φυσική, ιστορική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Ακόμη και γεωργική κληρονομιά. Επομένως, η οδή του Ίνου, Ιταλός είμαι, έλεος. Αν εγώ δεν εκτιμώ το, τις οδούς του Ίνου, αλίμονο. Όπως είπε και ένας άλλος συνάδελφος, υπάρχει και ένα σημαντικός θρησκευτικό τουρισμού. Σαντιάνκο Δικομποστέλα, Φερρυπίν. Αλλά όλη η Ευρώπη, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν τέτοιοι προορισμοί. Εγώ είμαι καθολικός, αλλά δεν μιλάω μόνο για τέτοιους καθολικούς α, τόπους. Α, ακόμα και μουσουλμανικοί και εβραϊκοί και χριστιανικοί αλλά μη καθολικοί τέτοιοι τόποι υπάρχουν. Γιατί μην ξεχνάμε, για το Ισλάμ θερυπή, μην ξεχνάμε τη σημαντική παρουσία του Ισλάμ στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να παρουσιάσουμε την Ευρώπη ε, ως ένα γενικό τουριστικό προορισμό. Ε, νομίζω ότι οι διάφορες θρησκείες ε, μπορούν να διαφοροποιήσουν και το είδος των τουριστών. Είναι πολύ σημαντικό για τις διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη, χάρη σε, μπορούμε να βρούμε διαδρομές για να συνδέσουμε διάφορες χώρες, από το βορρά μέχρι τον νότο της Ευρώπης. Και γι' αυτό που είπατε εσείς κυρία Μπιλμπάου, και η γεωργία ας πούμε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού. Ε, σκέφτομαι τον γαστρονομικό τουρισμό, αλλά και τον αγροτουρισμό, που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Πολλά άτομα ε, και όλο και περισσότερα θέλουν να, πάνε, να περάσουν τις διακοπές τους όχι στην παραλία, αλλά στην Ήπεθρο. Ε, και καλό είναι και για τα παιδιά μας, έτσι, τα οποία σε λίγο θα ξεχάσουν θα ξεχάσουν ε, πώς είναι τα ζώα. πούμε. Υπάρχουν παιδιά που δεν αναγνωρίζουν το γάιδαρο από το μουλάρι. Δεν ξέρουν, ας πούμε, τη διαφορά από το λαγό στο κουνέλι. Ε, στο κουνέλι. Καλό είναι να παίρνανε που και που, ας πούμε, τις διακοπές τους στην Ήπεθρο. Εγώ, ας πούμε, και τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά τα πήγαινα από εδώ και από εκεί για να τους ανοίξουν τα μάτια. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε στο πρώτο μας ραντεβού που έχουμε το Σεπτέμβριο. Θέλω να απαντήσω σε εσά, κύριε Μπάκ. Ήρθα σε επαφή με τη Γενική διεθνή του Συμβουλίου της Ευρώπης για να συζητήσουμε το θέμα των ποτιστικών διαδρομών. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν είναι κοινοτικό θεσμικό όργανο, ε, καλό να προωθηθεί, ε, γιατί μπορεί να προωθήσει και τα δικά μας θέματα. Ε, και μπορεί να βοηθηθεί η προσπάθεια αυτή χάρη στην υποστήριξη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Και στις 27 Σεπτεμβρίου που θα συζητήσουμε για τις θρησκευτικέ διαδρομές, ευκαιρία είναι να συζητήσουμε και την πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κύριε Φιδάνσα, μιλήσατε για την κινητικότητα στις πόλεις και τις προτάσεις της Κομισιόν για τα πιο καθαρά οχήματα. Κοιτάξτε, εγώ άλλαξα αρμοδιότητα, αλλά ο ίδιος άνθρωπος είμαι και επομένω τα αστικά θέματα, τα θέματα των πόλεων, δεν τα ξεχνάω και είναι η άλλη διάσταση τα θέματα των πόλεων στην ανακοίνωση που παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα για τα αυτοκίνητα που δεν μολύνουν τόσο. Τα αυτοκίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πόλεις μας, πόλεις που έχουν προβλήματα έντονα μόλυνσης. Τώρα, αυτή η στρατηγική βασίζεται σε δύο πυλώνες. Καταρχάς, ε, του κινητήρα καύσης ε, ούτω ώστε να, και, να μειώνονται όλο και περισσότερο οι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Επίση, ε, προωθεί μια στρατηγική μακροπρόθεσμη το υβριδικό αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και άλλα συστήματα ε, κινητήρων που λειτουργούν ψυχρό και που μολύνουν λιγότερο. Ε, η Ισπανική Προεδρία προωθεί πολύ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή και μπορούμε να την αναπτύξουμε. Ιδίως στο εσωτερικό των πόλεων, που υπάρχουν και προγράμματα από διάφορα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα. Τελευταίο θέμα, πριν να απαντήσω στον κύριο Σάβης, που αφορά και το παρελθόν μου, αλλά και το παρόν μου <laughs> ως επίτροπος. Μιλήσατε για την ε, επικουρικότητα και τις αρμοδιότητες των ε, περιφερειών. Υπάρχει αυτό το θέμα της επικουρικότητας με τα κράτη-μέλη. Ε, και υπάρχει και το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων των ε, διαφορών περιφερειών. Εγώ θέλω να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των τουριστών. Εγώ δεν αποφασίζω για την τουριστική πολιτική γενικά. Ξέρω ότι υπάρχουν εθνικές πολιτικές διαφορετικές και περιφερειακές τουριστικές πολιτικές πάλι διαφορετικές. Ε, υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμού. Δεν το αρνούμε εγώ αυτό. Εγώ θέλω να ενορχιστρώσω αυτές τις προσπάθειες σαν διευθυντής ορχήστρας. Ούτω ώστε όλες αυτές τις προσπάθειες να εναρμονίζονται οι μεν ε, με τις δε και να παραπλασιαστεί ο αριθμός των τουριστών. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, Μίλησα προηγουμένω για τη σημασία ε, του να έχουμε επαγγελματίε στον τομέα του τουρισμού. Έχει σημασία η κατάρτιση των επαγγελματιών, των νέων που δουλεύουν συχνά στον τομέα του τουρισμού. Ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, σχολέ που διδάσκουν τους νέους οι οποίοι ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα. Ε, που, είναι, που γίνονται διευθυντέ σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω να πολλαπλασιαστούν αυτέ οι σχολέ και αυτέ οι προσπάθειε στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να καταρτιστούν αυτά τα άτομα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε επίση και τα οικονομικά εργαλεία που έχουμε. Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την ε, επιχειρηματικότητα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και του νέου που ενδιαφέρονται για τα τουριστικά επαγγέλματα. Τώρα, το πρόβλημα των ε, ατόμων με, με μειωμένη κινητικότητα. Κάποιος στη Ματρίτη είπε ότι θέλω το δικαίωμα των ατόμων με κινητικά προβλήματα να το εξισώσω με το δικαίωμα στον τουρισμό. Θέλω δηλαδή, τι εννοώ, να επιτρέψω σε όλους όσους έχουν προβλήματα να υποφεληθούν ε, από την ομορφιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν μιλάω για μια, ένα δικαίωμα το οποίο θα γραφτεί μέσα σε μια συνθήκη και θα εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητας και που έχουν περισσότερες κοινωνικές δυσκολίες, καλό θα ήταν να έχουν τη δυνατότητα να ε, επισκεφτούν ε, ενδεχομένως σε περίοδους low season κάποιες τουριστικούς προορισμούς. Αυτό ε, ωφελεί και την οικονομία αλλά και την κοινωνική πολιτική. Γιατί όπως λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας, το, το βασικό μας εργαλείο είναι η αγορά. Αλλά η κοινωνική πολιτική είναι ο τελικός μας στόχος. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που ανέφερε η συνάδελφος από τη Βαλτική. Πολύ σωστά όσα είπατε. Όταν ήμουν επίτροπος μεταφορών το είχα συζητήσει με το συντονιστή που ασχολούνταν με τα δίκτυα. Υπάρχει ένα θέμα με τους σιδηροδρόμους. Η Ισπανία και η Πορτογαλία, το αντιμετωπίζουν ε, εδώ και πολλά χρόνια, δεν το έχουν επιλύσει ακόμα. Διάφορες χώρες που ανήκουν, ανήκαν στην Σοβιετική Αυτοκρατορία έχουν περισσότερα προβλήματα με τους σιδηροδρόμους από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι δύσκολο βεβαίω να φτάσει κανεί ορμικά στο Τάλιν. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια. Και σε μία από τι τελευταίε συναντήσει που είχα ω Επίτροπο Μεταφορών ε, ήταν να δεσμευτώ για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, βεβαίω τίθεται και ένα οικονομικό ζήτημα εδώ, έτσι, ε, σημαντικό. ελπίζω ο διάδοχός μου, κύριος Κάλλας, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος στα προβλήματα της βαλτικής περιοχής να βοηθήσει για να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που τον ενδιαφέρει έτσι και συναισθηματικά. Καλό θα ήταν ούτω ώστε όλες οι ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες να είναι προσπελάσιμες και συνδρομικά. Βέβαια εύκολα είναι τα λόγια, δύσκολες οι πράξεις, αλλά αν υπάρχει η δέσμευση και η πολιτική θέληση μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Thank you, Commissioner. Last round, I promise. We start with Mrs. Ε, δύο λεπτά. Α, ευχαριστώ, κύριε Πίτροπε, για την παρουσία σας σήμερα. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που υπόθηκαν. Επειδή ως Ευρωβουλευτής και ως υπευθύνη του τουρισμού στην πόλη μου, συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε. Είναι σημαντικό αυτός ο τομέας του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονιστεί σε πολλούς τομείς επειδή νομίζω ότι οι χώρες μας δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές λόγω του πλούτου που έχουν. Και προηγουμένως μιλήσαμε για όλες τις πολιτιστικές διαδρομές, για τον πολιτισμό, για τους αμπελώνες. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμπληρωματικά και νομίζω ότι στο δικό μου το επίπεδο το γαλλικό υπήρξαν κάποιες θέσεις ευθύνης και για τον επιχειρηματικό τουρισμό. Εγώ προσπάθησα να κάνω εναρμόνιση και να αποδείξουμε ότι αυτός ο επιχειρηματικός τουρισμός παραμένει σε μας στη Γαλλία σημαντικός και το ίδιο σε όλη την Ευρώπη γιατί αναπτύσσεται πολύ σημαντικά σε εμά σε σχέση με την ανάπτυξη του άλλες ε, υπήρους. Ελπίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε, εσείς και εμείς, όλοι μας δηλαδή, να έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά εργαλεία για να απτύξουμε αυτό τον ε, τουρισμό. Είπατε ότι η κατάρτιση είναι κάτι το σημαντικό. Εγώ όμως συνειδητοποίησα ότι είναι σημαντικό τα διαφορετικά ταμεία να βοηθούν όχι μόνο τις επαγγελματίε του τουρισμού, αλλά να διατηρούν και να προστατεύουν το, το, την πολιτιστική μας κοινωνία. Αυτά είχα να πω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τεκάλ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι όταν μιλάμε για τον κοινωνικό τουρισμό. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει κάποιες προκαταρκτικές δράσεις. Είμαστε στο δεύτερο έτος. Συντάσσουμε κάποιες μελέτες και 7 και 8 Μαΐου θα έχουμε μια διάσκεψη και τον Ιούνιο θα παρουσιαστούν μελέτες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κοινωνικό τουρισμό. Η Ισπανία έχει τέτοια έργα που συμπεριλαμβάνουν ένα εκατομμύριο ηλικιωμένους και το κράτος επενδύει 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αλλά εισπράττει 125 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Συμμετέχουν 500 ξενοδοχεία. Ο κοινωνικός τουρισμός στοχεύει σε φοιτητές, σε ανάπηρους και σε ηλικιωμένους. Θεωρώ πως ο κοινωνικός τουρισμός οδηγεί σε υψηλότερο αριθμό τουριστών σε περισσότερες ε, θέσεις εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε εάν ε, ε, σκέφτεστε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για αυτόν τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ κύριος Κουμουτσάκος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον ε, Επίτροπο κύριο Ταγιάννη. Επιτέλους κύριε Επίτροπο έχουμε νομική βάση για να κάνουμε τη δουλειά μας στον τουρισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ θετικό ότι όπως σας άκουσα ξεκινάτε δυναμικά, με όραμα και φιλοδοξία. Βεβαίως ταυτόχρονα με τον ενθουσιασμό σας βλέπω πολύ θετικά ότι υπάρχει και ρεαλισμός. Υπάρχει ένας συνδυασμός ενθουσιασμού και ρεαλισμού. Και ο ρεαλισμός έγκυται στο ότι επανελάβατε πολλές φορές ότι η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας θα είναι ένας σταθερός οδηγός των δραστηριοτήτων σας στην ανάπτυξη αυτού του πολύ σημαντικού τομέα δράσης για την ευρωπαϊκή οικονομία που είναι ο τουρισμός. Ε, από τις πολλές προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε δύο. Την ε, ανάγκη να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα βιωσιμότητα στον ευρωπαϊκό τουρισμό δηλαδή καλές τιμές αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί κύριε Επίτροπε ίσως θα έπρεπε να δούμε και να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επιβραβεύονται από την Επιτροπή συγκεκριμένες περιοχές σε κράτη-μέλη που έχουν σεβαστεί το περιβάλλον και είναι ταυτόχρονα έλξεως τουριστών. Αυτό θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στα κράτη-μέλη και να σέβονται το περιβάλλον και να έχουν μια συγκεκριμένη σταθερή πολιτική. Και η δεύτερη πρόκληση είναι πώς θα σεβαστείτε ταυτόχρονα την ανάγκη της προστιθέμενης αξίας ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για τον τουρισμό, αλλά και των εθνικών πολιτικών. Είναι πολύ θετικό ότι μιλήσατε για προστιθέμενη αξία. Το πιστεύω και εγώ, ότι η προβολή γενικά της Ευρώπης θα υπηρετήσει το συλλογικό συμφέρον των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής στο τέλος του χρόνου Πιστεύω κύριε Επίτροπε ότι για να έχει επιτυχία αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής διάλογος με το Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνταγή της επιτυχίας είναι διάλογος, διάλογος και διάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λιμπεράτσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και με την νέα σας ιδιότητα. θέλω να διαβάσω όλας ε, και την ομιλία σας, αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα τώρα για την τουριστική επέκταση μιας περιοχής απαιτούνται κάποια πράγματα όπως η πληροφόρηση, η διαφήμιση και βλέπουμε χώρες όπως η Ισπανία ή η Γαλλία που έχουν έντονη παρουσία και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ευρωπαϊκή ετικέτα όπως το είπατε η μάρκα Ευρώπη πράγματι πρέπει το να προσελκύσουμε τουρίστες εκτός Ευρώπης αλλά πόσες φορές μπορεί κανείς να πάει να δει τη Γαλλία και την Ισπανία γιατί όχι τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία ή τη Λιθουανία αλλά το πρόβλημα είναι πως δεν έχουν προωθηθεί αρκετά αυτές τις περιοχές και δεν έχουν αναπτυχθεί. Τώρα, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θεωρείτε εσείς πως μπορούν αυτά τα δύο μέσα να χρησιμοποιηθούν ένεργα μόνο 16% των ε, κονδυλίων αυτών των ε, προγραμμάτων ε, έχουν εκταμιευθεί. Θα μπορούσατε ίσως να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι προς την κατεύθυνση του τουρισμού. Για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, εύχομαι επιτυχία στα σχέδιά σας, αυτά τα οποία μας είπατε και μας είπαν οι συνάδελφοι μας έδειξαν ε, που μπορούμε να φτάσουμε να εργαστούμε σκληρά. Τρεις συγκεκριμένε σκέψεις ε, έχω να κάνω. Αναφέρατε και τις ε, τουριστικές σχολές. Εμείς στην Αυστρία έχουμε εξαίρετες για παγκόσμια γνώστες τέτοιες σχολές. Θα μπορούσε να υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ αυτών των σχολών των ευρωπαϊκών που θα βελτιώσουν την ποιότητα. Θα μπορούσαμε να το προωθήσουμε αυτό. Συγκεκριμένα τώρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί θα μπορούσε να είναι να ρυθμίσουμε τις διακοπές ε, έτσι ώστε να μην βγαίνουν όλοι μαζί στους δρόμους το καλοκαίρι. Αυτό θα βοηθούσε νομίζω και τον τουρισμό και θα ήταν και μεγάλη επιτυχία γιατί θα έφευγαν όλοι μαζί ταυτόχρονα ε, οι τουρίστες δηλαδή που θέλουν να πάνε στο ίδιο μέρος. Ξέρουμε εδώ πέρα τα ποτηλιαρίσματα στον αυτοκινητόδρομο κοντά σε μένα δεκάδων χιλιόμετρων για να μην μιλήσω καν για το τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Επίσης η Κομισιόν ε, έχει και τη σχετική οδηγία για τα ταξιδιωτικά πακέτα που βεβαίω είναι στην πλευρά της προστασίας των καταναλωτών και όχι του τουρισμού, ελπίζω να μπορέσετε να επηρεάσετε εδώ πέρα κάπως τα πράγματα. Και τέλος τα περιφερειακά προβλήματα και τα περιφερειακά έργα στον τουρισμό νομίζω πως έχουν ιδιαίτερη σημασία και προοπτική για το μέλλον. Ίσως και εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα ε, κάποιων ε, ενισχύσεων για να προχωρήσουμε. Κυρία Γκρίσμπεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Επίτροπο. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατη, αν και μερικές φορές ε, καθυστερώ. Ε, άκουσα τους στόχους σας, ε, τους προσυπογράφω. Ας επωφεληθούμε από αυτή τη θέλησή σας να γίνετε εσείς διευθυντής ορχήστρας ε, που θα παίξετε το δικό σας ρόλο ε, αρμονικά με τους υπόλοιπους ε, οργανοπαίκτες. Όπως είπατε, στον τουρισμό υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολλών θέσεων απασχόλησης. Είναι ο τρίτος οικονομικός τομέας, πάνω από 10% του εργατικού δυναμικού. Ας υποφεληθούμε για να αναπτύξουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική από κοινού όπου θα συμμετέχουν ε, διάφορες περιφέρειες και όπως είπε και η κυρία Βλαστό να χρησιμοποιήσουμε ε, και διάφορες ε, χρηματοδοτήσεις. Για το θέμα της χρηματοδότησης είναι κέρια σημασίας, κυρίως μέσω των διαφορετικών ταμείων για να απτύξουμε φερρυπίν τις περιφέρειες μέσω της χρήσης του ΦΕΑΝΤΕΡ να καταπολεμήσουμε την έξοδο από την Ήπεθρο, να φανταστούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε διάφορες θέσεις απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα. Κλείνοντας, η ιδέα σας για το, τη βιομηχανική ε, κληρονομιά μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ προέρχομαι από μια διασυνοριακή περιοχή, όπου αρχίζουμε αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την σιδηροδρομική βιομηχανική κληρονομιά. Θα μπορούσαμε να συνδεθούμε με το Λουξεμβούργο, τη ΣΑΡ, την Ανατολική Γαλλία, ε, σιδηροδρομικά. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Και φυσικά πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και τον τουρισμό των παιδιών. Καλό είναι να ξεκινήσουμε να εξηγούμε στα παιδιά κάποια πράγματα, γιατί ορισμένοι νομίζουν τα ραδίκια φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος. Να πω κι εγώ ένα-δύο πράγματα ως πρόεδρος. Η επικουρικότητα είναι πρόβλημα, γιατί τα κράτη, μάλλον οι βουλευτέ από την ε, Λετωνία, Εστονία, λένε και πώς θα έρθουν τουρίστες σε εμά. Οι Πολωνοί λένε πώς θα έρθουν ε, τουρίστες στην Πολωνία. Το πρόβλημα είναι θα έρθουν όταν προωθήσετε εσείς ε, τις ε, χώρες σας. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να λένε και θέλουμε και επικουρικότητα από τη μία και από την άλλη να λένε αλλά σας παρακαλώ μην κάνετε τίποτα ή μάλλον γιατί δεν κάνετε τίποτα για να προωθήσετε τη χώρα σας. Στη χώρα μου, ας πούμε, Προωθείται μόνο το Λονδίνο. Υπάρχει όμως και το Μάντσεστερ, Μάικλ. Αλλά οι τουρίστες που έρχονται στη Βρετανία πάνε μόνο στο Λονδίνο. Ε, στην, οι τουρίστες που πάνε στη Γαλλία πάνε στο Παρίσι, ε, στη Ρώμη, στην Ιταλία. Αυτό είναι το πρόβλημα της επικουρικότητας. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το πρόγραμμα ΕΔΕΝ, ε, προγράμματα αριστείας και η Βρετανική κυβέρνηση όμως αδιαφορεί πλήρως. Δεν θέλει να συμμετάσχει καθόλου σε αυτό το πρόγραμμα ΕΔΕΝ. Λόγω επικουρικότητας. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα με την επικουρικότητα. Αγαπητοί βουλευτές, δεν έχει νόημα να ρωτάμε την Κομισιόν τι θα κάνει για να βελτιώσει τον τουρισμό στην Λετωνία κτλ. Για στραφείτε σας παρακαλώ στις κυβερνήσεις σας για να τις ρωτήσετε τι θα κάνουν εν με τον τουρισμό εφόσον πριτανεύουν την αρχή της επικουρικότητας. Αχ, ωραία, το ξεφορτώθηκα αυτό το πρόβλημα. Τώρα, βιομηχανική κληρονομιά. Κύριε Επίτροπε, Ωραία ήταν αυτά που είπατε για τη βιομηχανική κληρονομιά. Πρέπει να αναπτύξουμε τη βιομηχανική κληρονομιά. Είναι η ιστορία της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο μάχες η ιστορία της Ευρώπης και οι μάχες με τα σπαθιά κτλ. Εδώ γεννήθηκε η βιομηχανική επανάσταση. Εδώ στην Ήπειρό μας. Είναι πολύ σημαντικό. Όλοι μας έχουμε βιομηχανική κληρονομιά. Καλό είναι να αναπτύξουμε. Όταν κοιτάμε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτεί και υποστηρίζει η Κομισιόν, υπάρχει μια προκατάληψη ε, για, για κάποια πούμε πολιτιστικά επιτεύγματα όπως η όπερα. Ε, δεν έχω πρόβλημα. Καλή είναι και η όπερα. Αλλά όταν βλέπουμε πώς, πώς πάνε τα χρήματα, πώς κατανέμονται, η όπερα βουτάει το 90% τη μερίδα του λέοντος από τα χρήματα. Έτσι, δεν είναι σωστό αυτό. Ε, και εδώ ε, συνδέουμε το ερώτημα της κυρίας Γκρίσμπακ για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε το βιομηχανικό ας πούμε, τουρισμό. Θα πρέπει να μοιράσουμε δίκαια την πίτα. Να μην τα δίνουμε όλα στα μπαλέτα και στην όπερα. Καλά είναι και αυτά βέβαια, αλλά όχι μόνο τα μπαλέτα. Ας το μοιράσουμε πιο σωστά αυτό το κέικ, αυτή την πίτα. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Βλέπετε αγαπητέ Επίτροπε, από την ποιότητα της συζήτησης, παρότι περιορίζονται οι βουλευτές ε, λόγω έλλειψης χρόνου, βλέπετε ότι και μόνο και μόνο τον αριθμό των ανθρώπων που πήραν το λόγο ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τον τουρισμό. Ε, για μας δεν είναι ε, δευτερεύον θέμα σε σχέση με τις μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικό σε με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους και περιμένουμε πραγματικά με ενδιαφέρον τη νέα σα ανακοίνωση και να είστε σίγουροι ότι θα σα υποστηρίξει αυτή η Επιτροπή για να αναπτύξετε μια πραγματική και ουσιαστική ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική υποστηρίζοντας διάφορα θέματα και προωθώντας και την το βιομηχανικό τουρισμό, τη βιομηχανική κληρονομιά. Αυτά που ζητήθηκαν θα τα κάνουμε. Όμω δυστυχώ βρισκόμαστε στην αρχή μια νέα φάση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό συλλέγοντας εμπειρίε του παρελθόντος αυτά δηλαδή που είχαν γίνει όταν ο τουρισμός δεν περιλάμβανε μια πραγματική νομική βάση τα πειράματα δηλαδή που έχει κάνει το κοινοβούλιο κλπ. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι είναι αποφασισμένη όπως και εγώ η Επιτροπή αυτή. Είπε και πρώτος ότι ο τουρισμός δεν είναι μια μεγάλη, μια από τις μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Αλλά νομίζω αυτό έχει αλλάξει και αυτό μας δίνει ελπίδα και η δική σας συμμετοχή στην συζήτηση με ιδέες, με προτάσεις αποδεικνύει ακριβώς ότι υπάρχει βούληση και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε σαφώς υπάρχει οικονομικό πρόβλημα αλλά βρισκόμαστε στην αρχή και όλες οι παλιές χρηματοοικονομικές προοπτικές δεν περιλάμβαναν τον τουρισμό ως τομέα κοινωτικής πολιτικής. Τώρα θα πρέπει μαζί να ξεκινήσουμε τη δουλειά ώστε τα κονδύλια από τον προπολογισμό για τον τουρισμό να είναι περισσότερα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Γιατί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σωστά χρησιμοποιώντας όπως είπε και ο κύριος Λιμπεράσκη και άλλα εργαλεία, διεθνωτικά ταμεία, Ευρωπαϊκό Τομείο Συνοχής κλπ. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και μια στρατηγική χρηματοοικονομική γιατί σωστά λέει ο κύριος Σίμψον να μην επικεντρωνόμαστε σε μία συγκεκριμένη κατάσταση μόνο γιατί υπάρχουν περισσότεροι τουρίστες οπότε πρέπει να διαφοροποιήσουμε και να κόψουμε καλύτερα την πίτα. Πριν όμως εγώ να αρχίσω να την κόβω την πίτα θα ήθελα να, μαγειρέψω, να τη μαγειρέψω καλά. Γιατί αν δεν είναι νόστιμη αυτή η πίτα είναι δύσκολο να την κόψουμε καλά. Προσπαθώντα έτσι να προωθήσουμε του διάφορου του τουρισμού. Και εγώ συμμερίζομαι με αυτό που είπε ο κύριο Σίμψον. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όμω και οι χώρε μέλη, όλε οι χώρε μέλη, να παίξουν και το δικό του ρόλο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο τουρισμό δεν είναι μόνο βασικό βασικός πόρος οικονομικός για τις χώρες του Νότου της Ευρώπης, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφθηκα τη Φιλανδία και σε συναντήσεις με την επιχειρηματική κοινότητα στο Ελσίνγκη άκουσα ότι και αυτοί έχουν θέληση να αναπτύξουν τουριστικά τη χώρα τους. Και η κυρία Πακ αναφέρθηκε στη σημασία του τουρισμού και για το Λουξεμβούργο. Δηλαδή, στο Μουσείο Τουρισμό είναι ένα πόρο για όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το σήμα αυτό το εμπορικό Ευρώπη να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να πω ότι όλοι οι υπουργοί τουρισμού που άκουσα στην ε, Μαδρίτη και αλλού και όλα αυτά που ακούσαμε σε σχέση για τις ε, ζημιές στον τουρισμό μετά από την σκόνη του φεστίου. Είδα λοιπόν να υπάρχει μια μεγάλη βούληση για δημιουργία ενός μεγάλου προγράμματος και καθησυχάστηκαν επειδή άκουσαν τη δική μου δέσμευση για μη επέμβαση στις αρμοδιότητες τους και επαναλαμβάνω, αυτή η συμφωνία Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, νομίζω μια πολύ καλή συμφωνία που κάλλιστα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλε χώρε και μάλιστα σα προσκαλώ τι υπόλοιπε χώρε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συμφωνία, ώστε να βρούμε πόρου και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Και ο κ. Τικάου νομίζω μίλησε, η κυρία Τικάου μίλησε για αυτό το θέμα της κοινωνικής συνοχής, του κοινωνικού τουρισμού, που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και μάλιστα επιφέρει και σημαντικά κέρδη. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της οδηγίας για τις αναρρές ε, μεταφορές κάλεσα να μου πω τη γνώμη τους δύο βουλευτές οι οποίοι μου είπαν ότι εντάξει πολύ καλά να έχουμε το δικαίωμα του ταξιδεύει αλλά πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στο αεροδρόμιο στη Λούρντ, στη Λούρδη, να δείτε πόσο κόσμο υπάρχει με μειωμένη κινητικότητα, να δείτε το, μεγάλο αριθμό τέτοιου, ε, τέτοιου είδους επιβατών που υπάρχει εκεί. Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε όταν μιλήσαμε προηγουμένω για τα δικαιώματα στον τουρισμό. Αλλά το ξαναλέω, ε, το δικαίωμα αυτό δεν είναι δικαίωμα που απορρέει από κάποια συνθήκη. Εμεί θα πρέπει πολιτικά να διασφαλίσουμε σε μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών που έχουν ε, κάποια ε, προβλήματα στην κινητικότητα να επιτρέπουν να να επιτρέψουν σε αυτού του ανθρώπου να ταξιδεύουν. Το πρόγραμμα το Ισπανικό ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα που είχε πολύ καλά αποτελέσματα με σημαντικά ε, οικονομικά κέρδη. Και για κάθε ευρώ που δαπανούσαμε κερδίσαμε 40 λεπτά. Αυτό θα πρέπει να το διευρύνουμε. Και θα πρέπει να διευρύνουμε επίση και την σεζόν. Να μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στον τουρισμό σε συγκεκριμένε περιόδου τη χρονιά, αλλά θα πρέπει να τι διευρύνουμε. Και εύχομαι για την Αυστρία που ασχολήθηκα τόσο όταν ήμουνα Επίτροπος Μεταφορών. Ελπίζω το πέρασμα στο Μπρένερο να επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των τουρισμών Πάντως θα προσπαθήσουμε να κατανείμουμε τις τουριστικές παρουσίες ε, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και να μην βασιζόμαστε μόνο στο high season. Συμφωνώ λοιπόν και με την ανάγκη διαλόγου γιατί η παρουσία μου εδώ δεν αποτελεί μόνο μια επίσημη παρουσία που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Εγώ ζήτησα να υπάρξει συμβολή συγκεκριμένη για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε και μάλιστα ξεκινήσαμε θα έλεγα από τις 9 του Φλεβάρι φέτος. Χρειαζόμαστε χρόνο βέβαια, χρειαζόμαστε σκέψη και συζήτηση και θα είμαι και στο Μαραθώνα στην εκδήλωση που οργανώνει η Ελλάδα για την ε, μάχη της Μαραθώνα σημαντικό αυτό γεγονός όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε να κάνουμε διάλογο και είμαι διαθέσιμος γι' αυτό. Και κάθε φορά που θέλει ο κύριος Σίμψον είμαι στη διάθεσή σας ε, να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και αναμένω από εσάς ενδείξεις, προτάσεις, συμβολές συγκεκριμένε, όσο δηλαδή εξελίσσεται η σύνταξη της ανακοίνωσης. Οι συναντήσεις που είχαμε ήταν ένα πρώτο ραντεβού, αλλά αυτά τα ραντεβού θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν στο μέλλον. Στο μέλλον. Βλέπω ότι ο χρόνος μου μειώνεται. Να πω και πάλι ότι είμαι απόλυτα δεσμευμένος στο να γίνει ο τομέας αυτός ένας τομέας ε, κινητήριας δύναμης της οικονομίας μας. Νομίζω ήδη η απάντηση που έχω ε, εκ μέρους του Κοινοβούλου είναι θετική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε πίτροπε και ελπίζω όταν θα πάτε στο Μαραθώνα αν προσπαθήσετε να μιμηθείτε τον Φιδιπίδη και να μεταφέρετε τα νέα της νίκης στην Αθήνα να μην έχετε καλύτερη μοίρα από τον Φιδιπίδη ο οποίος ε, όπως λέγεται είπε ναι νικήκαμε και ξέπνευσε. Ελπίζω όμως να εκτιμάει ο κόσμος την ιστορία και τη σημασία της μάχης του μαραθών ε, για την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού και την απόθεση των Περσών. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και για το ότι καθίσατε και πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις των συναδέλφων και ελπίζω να συνεργαστούμε στενά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. We'll have a minute Παραμείνετε για την συνεδρία.